συνάδελφοι, παρόλο που κάποιοι δεν έχουν φύγει από την αίθουσα, πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλά στην ημερήσια διάταξη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, ε, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, Εάν δεν υπάρξουν στάσεις αντιρρήσεις, εγκρίνεται χωρίς τροποποιήσεις. Σας παρακαλώ, χρειάζομαι ησυχία. Μπορείτε να κάνετε πηγαδάκια εκτός αιθούσης. Παρακαλώ, φύγετε από την αίθουσα. Σας παρακαλώ. Σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που φεύγετε. Αντίο σας. Σχεδόν τα καταφέραμε. Σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη. Αλλαγές στη γραμματεία της ΕΝΒΗ. Με χαρά να καλωσορίσω τον κύριο Φασίνα που άρχισε από την 1η Δεκεμβρίου να εργάζεται στην γραμματεία της ΕΝΒΗ από την DG Expo μας ήρθε και η κυρία Κανιεύσκε Νόιμαν ε, θα φύγει από τον Ιανουάριο από την Επιτροπή Ένβη. Τους ευχαριστώ και τους δύο για την συνεργασία τους ε, τα τελευταία χρόνια και τους εύχομαι από καρδιάς καλή τύχη. Ε, ευχαριστώ λοιπόν ε, για την διερμηνία. εστονικά, γελικά, δανέζικα και λετονικά δεν θα έχουμε. Η συνεδρία συμμεταδίδεται και ηλεκτρονικά με την εφαρμογή e-meeting και θα μεταδοθεί και στο διαδίκτυο. Σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη. Πάλι ψηφοφορία αλλά όσο κουρασμένοι κι αν είσαστε, είναι σύντομοι, θα τα κάνουμε γρήγορα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν μεταρρύθμιση για το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητής ο κ. Μπέλετ. Ξεκινάμε αμέσως με τη συμβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε. ψήφισαν άπαντες. Στα αλήθεια. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Ναι, με συγχωρείτε, παρασύρθηκα. Μισό, μισό λεπτό. Παραείστε αργοί. Πατήστε τα κουμπιά σας. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα ψηφίζουμε για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Πρόθεση των Πρωτοιμούχων Καλλιεργιών. Ο κύριος Χολβένη. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά κατά παρακαλώ να τα χέρια. αποχέ. ε, πρέπει να ελέγξω. 40 ελέγχουμε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Όχι, καταπίπτει. Α, ωραία. Το 50 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Αποχέ, απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά Αποχέ, απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχέ. Α, πρέπει να ελέγξουμε. 52. Πέρας. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. πέρας εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58. 58 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64, 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, 62 υπέρ, ελέγχουμε μάλλον. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξετε, να ελέγξουμε. Την 77. Πέρασε. Εγκρίνεται. σημαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 80. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ Α, την 93 να ελέγξουμε λοιπόν, την 93. Πέρας. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω το ΕΛΚ καθόλου. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά εποχές. απορρίπτεται 89 υπέρ κατά εποχές. εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 Α, καταπίπτει. 94 πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές να να ελέγξουμε το πρώτο με 94. Αλλά πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας. Πέρασε. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές. Δεν είμαι σίγουρος να ελέγξουμε. Θα βοηθούσε να σηκώνετε τα χέρια σας. Ξαναλέει ο πρόεδρος. Βοηθάει. Πέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά εποχές να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 100 πέρας εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτε, 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά πρέπει να ελέγξουμε την 106. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ αν θέλετε να ελέγξουμε την 118 παρακαλώ την 118 πέρας εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτω. 119 υπέρ κατά αποχές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 κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ηλεκτρονική ψήφος για το σύνολο. Πέρασε. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον συγητή και ευχαριστώ που μου θυμίζεται να ελέγχω. Λοιπόν, όσοι θέλετε να αποχωρήσετε για να πάτε να εορτάσετε, να το κάνετε αυτό με ταχύτητα και ησυχία.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 Show, okay. Uh, thank you and we will start immediately with our item 6 on our... Λοιπόν, το σημείο 6 τώρα της διατάξεως είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών ετήσια επισκόψης ανάπτυξη για το 2018. Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΕΛΚ, ο κύριος Μέλο. Ξυπνήστε κύριε, κύριε Μέλο, λέει ο πρόεδρος, γιατί έχετε και τον λόγο. Please, Let the Συνάδελφοι, αφήστε τον ε, εισηγητή να μιλήσει. Okay. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε στα πορτογαλικά. Η συζήτηση για το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι μια ευκαιρία για να δούμε τις δημοσιονομικές πολιτικές και τις πολιτικές για την οικονομία με ε, βασικό κριτήριο την βιώσιμη ανάπτυξη και εδώ προσπαθούμε με την έκθεση αυτή και σε συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές να δούμε πτυχές που θεωρούμε σημαντικές. Πρώτα απ' όλα αρχές που καθορίζονται μέσα από τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, κοινή ευθύνη των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μια πρόκληση αλλά μαζί και ευκαιρία, ο τομέας της υγείας που θεωρείται μια αξία αυτή καθεαυτή, ο τομέας της υγείας μπορεί να προσφέρει κέρδος για την οικονομική ευημερία και την κοινωνική συνοχή και στην περίπτωση αυτή, στη συγκεκριμένη συγκυρία, μας ενδιαφέρει και ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας για να δημιουργηθεί και ένα απόθεμα ιδίων πόρων που να συμπληρώνει τους εθνικούς και να ενισχύουμε τη δυνατότητα συλλογικής απόκρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάτι που θα επιτρέψει να ε, προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε δασικές πυρκαγιές και ούτω καθεξής. Η ξηρασία ε, στη Νότιο Ευρώπη άλλες φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, όλα αυτά απαιτούν να ε, επιδιώξουμε ακόμη περισσότερο την επίτευξη των στόχων που θέσαμε στη Συμφωνία των Παρισίων. Επίσης, θέλουμε μια στρατηγική προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης για τα δάση μας, για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Αυτά εν ολίγης, ε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτήν την εισήγηση. Δεν βλέπω άλλους σκιώδεις από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Από την Κούε, κυρία Κονέτσινα, δεν είναι εδώ. Υπάρχει κανείς που να θέλει το λόγο μεταξύ των συναδέλφων. Όχι, οπότε λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μ' ακούτε, διότι δεν βλέπω το μικρόφωνο μου. Αλλά το κοινοβούλιο μάλλον έχει ξεχωριστεί τόσο πολύ που μ' ακούτε. Σας παρακολουθούν όλοι σε όλα τα γραφεία, ξέρετε. Γεια σας. Είμαι διευθυντής υπεύθυνος για την εκτέλεση και την στήριξη προς τα κατημέλη στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει την Επιτροπή ΕΝΒΗ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξή της και που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, με την παραβολωτική διάσταση της ετήσιας έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο της ετήσιας επισκόπησης και ε, θέλουμε όντως περισσότερο πρασίνισμα της ετήσιας επισκόπησης και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έχουμε μια σειρά από σχόλια από, την, από το σχέδιο γνωμοδότησής σας στην ε, παράγραφο 1. Το σχέδιο έκθεση ζητά ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις και τις επιλεκτικές επενδύσεις με επενδύσεις σε τραγικές περιοχές θα είδατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στις 22 Μαΐου φέτος δήλωνε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και στόχοι της τώρα περιλαμβάνονται πλήρως στο εξάμεινο. Η ετήσια επισκόπηση για το 2018 ε, για την ανάπτυξη επικεντρώνεται περισσότερο στην βιώσιμη ανάπτυξη Εκεί δηλώνεται ότι οι επενδύσεις που θα, θα προωθήσουν την περιβαλλοντική ε, βιωσιμότητα και μπορεί να ενισχύσουν την πραγματικότητα όλη τη οικονομία με την καλύτερη διαχείριση των πόρων και τη μείωση της κατασπατάλησης πόρων και κόστους και του εξωτερικού κόστους και αντικτύπου θα ε, προτιμηθούν. Επίσης, η ανακοίνωση τονίζει ότι οι επενδύσεις σε τομείς όπως η υγεία και η κυκλική οικονομία μπορεί να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την απασχόληση. Οι δημόσιες προμήθειες, οι επενδύσεις, τη διαχείριση των υδάτων και των ε, ε, αποβλήτων. Η χρήση βιοκαυσίμων και βιοχημικών είναι συγκεκριμένα παραδείγματα τον οποίο πρέπει να εργαστούμε. Θα, θα, θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε από την Επιτροπή ΕΝΒΗ να μας υποστηρίξει. Να ε, συμπεριλάβει μια μνήα και στους τομείς αυτούς. Στην παράγραφο 8 του σχεδίου έκθεσης καλείται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει μια βιώσιμη στρατηγική για τα δάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί απολύτω για την σημασία τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και τη δασοκομεία και την ανάγκη τα δάση όχι απλώ να γίνουν πιο ανθεκτικά στι συνέπειε των κλιματικών αλλαγών, αλλά να χρησιμοποιηθούν καλύτερα και οι δυνατότητέ του για να αναχαιτήσουμε τον αντίκτυπο των κλιματικών αλλαγών και να χρησιμοποιηθούν ω ε, καταβόθρε άνθρακα με σημεία αποθήκευσης άνθρακα. Η νέα στρατηγική για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές λοιπόν μπορεί να το λάβει υπόψη αυτό ε, και άλλα νομοθετικά εργαλεία μας διατίθενται για να στηρίξουμε αυτά τα στοιχεία, η οδηγία Nature, τα κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία, η κοινή αγροτική πολιτική και το καθεξής. Ε, πολύ πρόσφατα, στις 23 Νοεμβρίου 2017, με, με την ε, πρικαγιές ε, στην Νότια Ευρώπη και γενικότερα τον κίνδυνο από τις κλιματικές αλλαγές, προτείναμε τη δημιουργία ενός νέου αποθεματικού ως μέρος ε, του συνολικής δυνατότητας ε, πολιτικής προστασίας και για την... Ε, δυνατότητα απόκριση σε ξαφνικέ φυσικέ καταστροφέ όπω τι δασικέ πυρκαγιέ. Βασικέ προκλήσει όλων αυτών των στόχων και πολιτικών και τη πρακτική του υλοποίηση είναι κάτι που πρέπει να το προωθήσουμε και χάρη στη δική σα έκκληση για την καλύτερη διαχείριση των δασών και τη δασοκομεία. Στην ουσία δηλαδή τα σχόλιά μα είναι σε δύο επίπεδα. Συμφωνούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΕΝΒΗ να υποστηρίξουμε τη συμπερίληψη πιο συγκεκριμένων τομέων, όπως λέει η παράγραφος 1 του σχεδίου έκθεσης. Και το δεύτερο σχόλιο μας έχει να κάνει με τις προτάσεις σας για τα δάση. Τις καλωσορίζουμε θερμά. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας. Λοιπόν, είδα κάποιον ε, άλλον από την Κομισιό ε, που έχει ζητήσει το λόγο επίσης. Ναι. Ωραία. Σύντομα. Ναι. Πολύ σύντομα. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή σας εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα. Παρακολουθούμε τις έργες σας, το έργο σας, τις απόψεις σας. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο βέβαια είναι μια δυναμική διαδικασία και απλά ήθελα να σας πω ότι είμαστε ανοιχτοί και σε μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ της δεν θέλει να ξαναλάβει το λόγο. Οπότε, 13 Δεκεμβρίου στις 11 το μεσημέρι είναι η προθεσμία καταβολής τροποθεσμών. 23-25 Ιανουαρίου θα γίνει η ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ. 22 Φεβρουαρίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. αυτά. Να δω αν, έχουμε, αν είναι εδώ ήδη οι προσκεκλημένοι μας προκειμένου να να συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα της εμείς διάταξης. Μάλλον πρέπει να περιμένουμε τον κύριο Ράζι να καταφτάσει. Um, uh, Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 7. Ετήσια ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Κουίντο Ράζη, εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, στο πλαίσιο του τακτικού διαλόγου που έχουμε με τον EMA. Χαιρόμαστε λοιπόν που έχουμε την ε, δυνατότητα να συζητήσουμε σήμερα μαζί του το πρόγραμμα εργασιών 17-18 υπό τη σκιά των εξελίξεων ε, που υπήρξαν σε κάποια κράτη-μέλη. Μας πείτε τι έχει συμβεί. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, καλημέρα. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα για άλλη μια φορά να λογοδοτήσω για το τι κάναμε την προηγούμενη χρονιά. Και θέλω να δράξω αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την κυρία Μπιλιάνα Μπόρζα για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε μαζί της. Λοιπόν, έπειτα από πάνω από ένα ολόκληρο έτος φοβερή αβεβαιότητα. Ένα στοιχείο αυτή τη αβεβαιότητα τουλάχιστον έχει εκλείψει. Γνωρίζουμε πλέον ότι μετακομίζουμε στο Άμστερνταμ. Η μετακόμιση του οργανισμού και η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φαρμάκων εν ώψη της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί τεράστια ποιήση στις δραστηριότητε μας. Ήδη πάνω από 40 μέλη του προσωπικού μας ε, εργάζονται αποκλειστικά επ' αυτού και φυσικά ως εκ τούτου δεν είναι διαθέσιμοι να εκτελέσουν τα κανονικά τους ε, καθήκοντα. Και όλα αυτά προστίθενται στις περικοπές προσωπικού που αναγκαστήκαμε να κάνουμε τα τελευταία πέντε χρόνια παρά το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρή και σταθερή αύξηση, αύξηση του φόρτου εργασίας μας και του προϋπολογισμού μας. Γι' αυτό και είμαι βέβαιος ότι δεν σας εκπλήσει το ότι θα σας πω ότι πολλές από τις δραστηριότητε μας έχουν ήδη πληγεί και επηρεαστεί από την κατάσταση αυτή. Εσωτερικά έχουμε περικόψει εκπαιδεύσεις, ελέγχους, χρειάστηκε να καθυστερήσουμε μια αναγκαία αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής μας, γιατί χρειάστηκε να δώσουμε προτεραιότητα ε, στα έργα ε, τηλεματικής ε, σε ενωσιακό επίπεδο και βεβαίως ε, χρειάζεται πλέον να επικεντρωθούμε και στην φυσική μετατόπιση, με την κατάσταση των υποδομών μας. Εξωτερικά χρειάστηκε να μειώσουμε την ταχύτητα με την οποία θέτουμε στη διάθεση του κοινού τα δεδομένα κλινικών δοκιμών, βάσει των οποίων βγάζουμε εμεί τι συστάσεις μας. Χρειάστηκε να μειώσουμε σοβα, σημαντικά τον αριθμό συναντήσεων και συνδιασκέψεων με μπυλακόμενους φορεί και εταίρους και χρειάστηκε να αναστείλουμε τα σχέδιά μας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πόρταλ με δημόσιες πληροφορίε για όλα τα φάρμακα που έχουν ε, άδεια κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεχομένως ε, μέχρι στιγμής κανείς να μην, να μην έχει παρατηρήσει ε, αυτές τις ε, αλλαγές λόγω του γεγονότο ότι το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ανταποκρίνονται στο 100% των δυνατοτήτων τους και προσπαθούν να μην μείνουμε πίσω σε τίποτα. Όμως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι διότι στο μέλλον ε, ο αντίκτυπος στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων μας προφανώς και θα γίνει <coughs> ορατός αναπόφευκτα. Έχοντας όλα αυτά κατά νου λοιπόν, ε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο φέτος γιατί παρόλα όσα αντιμετωπίσαμε καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις βασικές μας ευθύνες και μάλιστα στο επίπεδο το, της ποιότητας που γνωρίζετε από εμάς. Και πρέπει επίσης να σας ενημερώσω και για κάποιες πρόσθετες δραστηριότητες που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε πριν που μπούμε βέβαια σε αυτή τη μεταβατική φάση. Για παράδειγμα, πριν από δύο εβδομάδες βγήκε στον αέρα ένα νέο και βελτιωμένο σύστημα Udra Vigilance. Είναι ένα σύστημα ενημέρωσης που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για την υποβολή εκθέσεων σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες για παρενέργειες ορισμένων φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το νέο εργαλείο καθιστά την ενημέρωση και την ανάλυση των πληροφοριών αυτών πολύ πιο εύκολη. Κάτι που θα βελτιώσει την ασφάλεια των ασθενών. Το Σεπτέμβριο επίσης διοργανώσαμε την πρώτη μας ακρόαση στον EMA και η συνάδελφός σας, η Λίντα Μάκβαν, δήλωσε στην δημοσιαυτή Ακροασία το να δώσει κανείς στους ασθενείς μια πλατφόρμα για να πούν τη δική τους πλευρά, τη δική τους ιστορία, είναι αυτό που πρέπει κανείς να κάνει. Και θέλω να συμφωνήσω μαζί της και να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή την ε, Επιτροπή ΕΝΒΗ για το γεγονός ότι ήσασταν καθοριστική σημασίας ε, ε, εταίροι για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε αυτή την δημόσια ακρόαση. Επίσης, αυξήσαμε τις προσπάθειές μας για την άμεση συμμετοχή με τους κατασκευαστές, τους παραγωγούς για την δημιουργία καλύτερων ε, στοιχείων. Μάλιστα, σπάσαμε κάθε ρεκόρ το 2017 όσον αφορά τις επιστημονικές μας συμβουλές και αυτές οι διαδικασίες όλο και περισσότερο συμπεριλαμβάνουν ε, τους ασθενείς αλλά και φορείς αξιολόγησης ε, τεχνολογίας υγείας. Όλα αυτά τα επιτεύγματα λοιπόν που σας παρουσιάζω μας ε, θέτουν σε ένα καλό σημείο καθώς ε, εισερχόμαστε τώρα σε αυτήν την 16μηνη μεταβατική περίοδο για τη μετακατάστασή μας στο Άμστερνταμ. Βεβαίως η πόλη αυτή ε, έχει πολλά θετικά στοιχεία, είναι πολύ καλά συνδεδεμένη και η μεγάλη πλειοψηφία του προσωπικού του EMA έχει δηλώσει ότι είναι πιθανό να μετακομίσει στο Άμστερνταμ, να μα ακολουθήσει δηλαδή. Αλλά πρέπει να είναι σαφέ. το να μετακινήσει έναν τόσο μεγάλο οργανισμό όπω είναι ο EMA σε μια νέα χώρα είναι τουλάχιστον στην καλύτερη των περιπτώσεων πάρα πολύ περίπλοκη διαδικασία. Βεβαίω όλη αυτή η διαδικασία έχει, έχει καταστεί ακόμη πιο δύσκολη λόγω του φιλόδοξου χρονοδιαγράμματος καθώς θα πρέπει να έχουμε καταλήψει Λονδίνο το Μάρτιο του 2019. Είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά υπάρχουν πολλά εμπόδια που πρέπει να υπερπηδήσουμε. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουμε είναι ότι κατά το χρόνο που θα χρειαστεί να μετακομίσουμε, το νέο κτίριό μας στο Άμστερνταμ δεν θα είναι έτοιμο. Βεβαίω συνεργαζόμαστε με την Ολλανδική κυβέρνηση για να βρούμε μια ε, κατάλληλη ενδιάμεση λύση και αυτό το θέμα πρέπει να διευθετηθεί γρήγορα, διότι το ενδιάμεσο αυτό κτίριο θα είναι κρίσιμη σημασία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τι δραστηριότητέ μα από το Μάρτιο του 19 και έπειτα. Η άλλη μεγάλη μεταβλητή είναι πόσοι από, τελικά πόσοι από, τους, από τα μέλη του προσωπικού μας θα μας ακολουθήσουν στο Άμστερνταμ. Οι εσωτερικές μας εκθέσεις έχουν δείξει ότι έως και το 81% του προσωπικού μας θεωρεί πιθανό να μετακινηθεί, αλλά αυτό είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση ένας στους πέντε ε, εργαζόμενούς μας δεν θα μας ακολουθήσει. Σχεδόν 200 άνθρωποι δηλαδή. Και αυτή η απώλεια αυτού του μεγέθους μάλιστα προφανώς και θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις μας, τις δραστηριότητες μας και επιπλέον δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος ακριβώς θα έρθει, ποιος θα, ποιος θα μετακομίσει στο Άμστερνταμ, άρα δεν ξέρουμε και ποιο είναι το είδος των γνώσεων και της εμπειρογνωμοσύνης που μπορεί να χάσουμε. Και αν λάβει κανείς υπόψη ε, πόσο βαθιά εμπειρογνωμοσύνη και γνώση χρειάζεται κανείς για να δουλεύει στον EMA, η κάλυψη αυτού του κενού μπορεί να ε, πάρει πολλά χρόνια. Επίσης, έχουμε κάνει σχεδιασμό για το δίκτυο. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου σημαίνει προφανώς ότι το, ο φόρτος εργασίας μας θα πρέπει να ανακατανεμηθεί στους 27. Ε, Την ε, προηγούμενη χρονιά λοιπόν έχουμε ήδη κάνει κάποια ανάλυση προκειμένου να προσδιορίσουμε πιθανά κενά στην εμπειρογνωμοσύνη που θα χρειαστεί να ε, αντιμετωπίσουμε. Και πρέπει βεβαίω να σας πω ότι ε, μας ε, δίνει θάρρος η προδραστική προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει πολλά κράτη-μέλη, γιατί πολλά από αυτά έχουν ήδη λάβει συγκεκριμένα μέτρα και επενδυτικά και ως προς τις προσλήψεις προσωπικού, προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό που θα δημιουργήσει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Με τις κοινέ μας προσπάθειες λοιπόν του EMA και των κρατών μελών, θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε τουλάχιστον τις βασικές μας δραστηριότητες, βεβαίως χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστούμε. Θα επηρεαστούμε στους εξή τομεί, Ε, εκπαιδεύσεις, έλεγχοι, ε, συζητήσεις με εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης, θα χρειαστεί να αναβάλουμε ή να επιβραδύνουμε την εφαρμογή συγκεκριμένων νομοθετικών νομικών πράξεων, όπως είναι ο κανονισμός για τα κτηνιατρικά, η οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Θα χρειαστεί επίση να καθυστερήσουμε την εφαρμογή του σχεδίου δράση για, για τα φάρμακα προηγμένη θεραπεία και θα χρειαστεί να καθυστερήσουμε και τη συνεργασία μα με, με την διαμεσολαβήτρια στο τέλος, στο τομέα μάλλον της άμεσης ε, συμμετοχής. Και αυτό είναι πραγματικά μεγάλη απογοήτευση για μας γιατί είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και ε, πολύ θετική ε, επίδραση της, ε, της δραστηριότητας της κυρίας Οράιλη στο, στις διοικητικές μας πρακτικές. Η πρόσφατη μάλιστα θετική άποψη, γνωμοδότησή της για το έργο μας στον τομέα των εμβολίων για το HPV ήταν ένα από τα παραδείγματα για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την δημόσια εμπιστοσύνη στο έργο μας. Κύριε Πρόεδρε, ε, βρισκόμαστε σε ένα στο σημαντικότερο σταυροδρόμι για τον EMA στην 22χρονη πορεία του. Με την επιλογή του Άμστερνταμ μπορούμε ευλόγως να περιμένουμε ότι δεν θα υπάρξει κρίση στη δημόσια υγεία, δεν θα υπάρξουν ελλείψεις στην παρακολούθηση της ασφάλειας φαρμάκων, ούτε σημαντικές καθυστερήσεις στην έγκριση νέων φαρμάκων. Ωστόσο, το τίμημα ε, θα χρειαστεί να το πληρώσουμε σε πολλούς άλλους τομείς όπως σας εξήγησα. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μια έκκληση προς εσάς. Αντιμετωπίζουμε μια τεράστια πρόκληση μπροστά μας και μπορούμε να, την, ε, να ανταποκριθούμε σε αυτήν μόνο με τη δική σας διαρκή υποστήριξη. Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Καβεθόν Ρουίθ που θα μιλήσει εκ μέρους του υπευθύνου επαφής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, διευθυντή του οργανισμού. Αντιλαμβάνομαι απολύτως τις δυσκολίες που πάντοτε μια τέτοια αλλαγή ενέχει. Και έγινε προφανώς μια προσπάθεια ώστε αυτή η μετάβαση να είναι ομαλή και υποφελής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ από πλευράς μου είχα εκφράσει την προτίμηση προς την ε, Βαρκελόνη, αλλά βέβαια αντιλαμβάνομαι και το γενικότερο πλαίσιο που είμαι βέβαιο ότι θα ε, επιληθεί. Τώρα, ένα θέμα που ήθελα να θέσω ήταν το θέμα των εμβολιάσεων και των ε, κινήτρων για την έρευνα ο ΕΜΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτού ε, έχει αναλάβει τις ε, κεντρικές αδειοδοτήσεις για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που θεωρούνται ειδική ε, χρήσεως αλλά και των ορφανών τα οποία εν πάση σήμερα δυσκολεύουν την πρόσβαση των διαφόρων κρατών μελών προκειμένου να έχουμε καθορισμένη τιμή και αποζημίωση για τους πολίτες. Και έχουμε και φάρμακα τα οποία είναι όλο και πιο εξειδικευμένη χρήσεως. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα κινήτρων για την προώθηση των φαρμάκων αυτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως μια φαρμακευτική τάση, ίσως όχι βραχυπρόθεσμη αλλά μακροπρόθεσμη, όπου σημαίνει ότι οι ομάδες στόχου είναι όλο και πιο μικρές και η έρευνα αλλάζει στοχεύσεις. Αυτά τα κίνητρα λοιπόν ε, αναθεωρούνται και θα πρέπει να αναθεωρηθούν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να είναι οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη η χρήση αυτή. γιατί θα πρέπει να μπορέσουμε να προσφέρουμε τα κίνητρα αυτά, αλλά όχι μόνο να είναι αυτά τα προϊόντα προσβάσιμα για, την, για τους πολίτες. Και δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά με τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν, αν πρέπει να είναι το σύνολό τους και σε ποιους θα πρέπει να δίδονται. Και το λέγω αυτό στο πλαίσιο που συζητούμε για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και ιδιαίτερα αναθεωρώντας ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί προς το, ζήτημα της ε, μικροβιακής αντοχής. Και επίσης πώς βλέπετε σε μέσο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο το θέμα των ε, πιστοποιητικών αποκλειστικής εμπορίας για τα εμβόλια. Τα χρειαζόμαστε, αλλά ανησυχώ σχετικά με την χρησιμοποίηση και την εκστρατεία που γίνεται σε πολλά μέρη της Ευρώπης σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους ε, υποβάλλονται ομάδες του πληθυσμού σχετικά με τους εμβολιασμούς που χρειάζονται. Νομίζω ότι θα ήταν απαραίτητη λοιπόν μια εκστρατεία ενημέρωσης για τους πραγματικούς κινδύνους που ενέχουν οι εμβολιασμοί αυτοί, ώστε να έχουμε επαρκής εγγύησης προς τους πολίτες και να αντιμετωπίσουμε τις τάσεις αυτές οι οποίες εν τέλει θα έχουν αρνητική επίπτωση επί των πολιτών. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ράζη. Κατανοώ βεβαίως ότι η μετακόμιση από το Λονδίνο στο Άμστερνταμ είναι ένα θέμα που σας απασχολεί. Άλλωστε, το είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά αυτό το θέμα πριν από λίγους μήνες. Είχα πει τότε ότι θα πρέπει η πόλη ε, στην οποία θα μετακομίσετε να είναι κατάλληλη ε, και ότι δεν, δεν πληρεί βεβαίω ε, τα κριτήρια αυτά η κάθε πόλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν λοιπόν πολύ θετικό το γεγονός ότι επελέγει το Άμστερνταμ. Είναι προφανές λοιπόν ότι χρειάζεται να, να διαθέσετε πολύ προσωπικό για αυτήν την μεταγκατάσταση. Αλλά συγχωρήστε με, το να, μιλάτε, το να έρχεστε εδώ και να μιλάτε μόνο για ε, τη μεταγκατάστασή σας, αυτό είναι απαράδεκτο. Ε, θα μπορούσαμε, αν θέλετε, να μιλήσουμε όλη μέρα και για το Brexit, αλλά οι πολίτες περιμένουν πολύ περισσότερα από εμάς. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε συγκεκριμένες πολιτικές προτεραιότητες και να ε, επιλύουμε συγκεκριμένα προβλήματα, καθώς αυτά ανακύπτουν. Και το ίδιο περιμένω και από τον EMA και το προσωπικό του. Η κυρία Καμπεσόν αναφέρθηκε σε ορισμένα ζητήματα που μας απασχολούν. Και θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω μαζί της. Πέρα από το Brexit υπάρχουν και τα προβλήματα της δημόσιας υγείας και των φαρμάκων. Και θέλω να τοποθετηθείτε για ένα συγκεκριμένο θέμα που μας απασχολεί. Η μικροβιακή εντοχή. Έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό πολύ συχνά και όπως σας έχω ξαναπεί, δεν είναι δυνατόν να μιλούμε μόνο για αυτό το θέμα και ποτέ να μην αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες δράσεις. Το Κοινοβούλιο έχει καλέσει πολλές φορές την ε, Επιτροπή να βοηθήσει και να διευκολύνει τη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου συστήματος για την ε, παραγωγή νέων αντιβιωτικών. Δεν είναι εύκολο το θέμα, ούτε θέλω να υπονοήσω κάτι τέτοιο, αλλά είναι αναγκαίο. Σχετίζεται το θέμα αυτό με την ποιότητα των αντιβιωτικών, με την χρήση των ε, αντιβιωτικών, διότι αν δεν κάνουμε ε, αυτό θα ε, καταλήξουμε να έχουμε παθογόνους μικροοργανισμούς οι οποίοι θα είναι αθάνατοι, που δεν θα μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό και τα επόμενα χρόνια χρειάζεται τα αντιβιωτικά να ρυθμίζονται με πάρα πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Εγώ μίλησα μάλιστα και προσωπικά με τον Ζαν Κλοντ Γιούγκερ ο οποίος με ενημέρωσε ότι δεν προτίθεται η Κομισιόν να υποβάλει καμία νομοθετική πρόταση. Και μάλιστα έως τον Ιούνιο του επόμενου ε, χρόνου θα υποβάλει τις τελευταίες νομοθετικές προτάσεις από τον Ιούνιο του 2018 καμία άλλη. Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα τρία χρόνια δεν θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Και εδώ θέλω συγκεκριμένη και σαφή δήλωση από τον EMA. Έχουμε τρία χρόνια στη διάθεσή μα. Μπορούμε να περιμένουμε οι, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί να γίνουν τόσο δυνατοί και τόσο ανθεκτικοί ώστε να πεθαίνει κόσμο στα νοσοκομεία μα Ή μήπω θα έπρεπε και εσείς να μα υποστηρίξετε και να μα πείτε ότι χρειαζόμαστε άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να ρυθμίζεται η χρήση και η ποιότητα των αντιβιωτικών, διότι είναι σαφέ. Είναι σοβαρό το θέμα. Πεθαίνουν άνθρωποι και εμεί καθόμαστε και συζητούμε περί ανέμων και υδάτων και μάλιστα δεν έχουμε και συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία επί της οποίας ε, να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε κυρία Ντάλη. Ευχαριστούμε καθηγητά Ράζη που είστε εδώ για να μας ενημερώσετε για όσα συμβαίνουν για την ε, μετακόμιση. Καταλαβαίνω ότι είναι τεράστια δουλειά και ακόμη πιο ε, δύσκολη γίνεται λόγω και της πίεσης χρόνου. Κάποια στιγμή Μιλήσατε και για την περίπτωση να μην υπάρχει ενδεχομένω ένα κτίριο ε, στο Άμστερνταμ όπου υποχρεώσετε να μετακομίσετε σε πρώτη φάση και δεδομένη τέλο πάντων αυτής της μετακίνησης που είναι κάτι το δύσκολο και τη σοβαρή δουλειά που έχει να κάνει ο οργανισμό σα για ένα σωρό θέματα, καταλαβαίνουμε πόσο λεπτό γίνεται το όλο ζήτημα. Όμω, ήθελα να μου πείτε, εάν έχετε ήδη επεξεργαστεί ένα ενδεχόμενο εναλλακτικό σενάριο. Εάν δεν μπορέσει να γίνει η μετακόμιση σε ένα κτίριο στο Άμστερνταμ εντό τη ημερομηνία όπου θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και πώς το σκέφτεστε αυτό. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερες πληροφορίες, πέραν όμως της μετακόμισης. Αυτό είναι προφανώς λεπτό, εξαιρετικά λεπτό θέμα, αλλά θέλω να σας θέσω κι εγώ μια σειρά από ερωτήσεις που ε, προφανώς εξετάζετε εσείς ως οργανισμός. Αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος ήδη, η αντίσταση στα αντιβιωτικά. Ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας ως Επιτροπή και προφανώς για όλο το Κοινοβούλιο. Είναι ένα θέμα που μας ανησυχεί. Όλοι συζητούμε με διαφορετικούς εμπειρογνώμονες και ε, επαγγελματίες που έχουν να μας πούν περισσότερες πληροφορίες εκ των έσω για τα διάφορα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι. Αλλά αν δούμε και τα στατιστικά στοιχεία, καταλαβαίνετε την έκταση του θέματος. Ε, καταλαβαίνετε ότι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στηρίζει, στοιχίζει 1,5 δις ευρώ η αντίσταση στα αντιβιωτικά. Κάτι που δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Και τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, λένε τα στοιχεία ότι οι ε, ασθένειες λόγω της αντιμικροβιακής αντίστασης μέχρι το 2050 θα προκαλούν ε, πάρα πολλούς θανάτους, ήταν η πρώτη πηγή και επίσης προκαλούν 25.000 θανάτους ετησίως. Ε, καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό θέμα είναι η αντιμικροβιακή αντίσταση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Ε, ιδίως τι κάνετε για να πάρετε πληροφορίες από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που είναι η βασική πηγή και τους γιατρούς που είναι αυτοί που κατεξοχήν συνταγογραφούν τα αντιβιωτικά. Τι κάνετε λοιπόν για την στρατηγική αυτή, για την αντιμικροβιακή αντίσταση και τα αντιβιωτικά στην ε, πολιτική δημόσια και για τις κλινικές δοκιμές και τη σχετική πολιτική. Αυτή ε, συμφωνήθηκε το 2014. Αλλά σκοπεύουμε να τεθεί σε ισχύ διότι ο οργανισμός ε, θα δημιουργήσει μια νέα βάση δεδομένων, ε, υποτίθεται. Θεωρείται ο κανονισμός αυτός πολύ σημαντικός, διότι θα πρέπει να παροτρύνει τη νέα έρευνα, αλλά και να διασφαλίσει την διαφάνεια στα αποτελέσματα των δοκιμών θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε σε τι φάση βρίσκεστε σε σχέση με την υλοποίηση του κανονισμού, με το τι πρέπει να περιμένουμε και με το ενδεχόμενο χρονοδιάγραμμα για το πότε αυτή η βάση δεδομένων μπορεί να έχει περατωθεί. Και μια τελευταία ερώτηση για την αναμενόμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τεχνολογίες της ε, αποτίμησης της υγείας. Βλέπω ότι ο οργανισμός των φαρμάκων έχει ρόλο να διαδραματίσει στην προετοιμασία μέσα της πρότασης, αλλά με απασχολεί κατά πόσον βλέπετε εσείς ένα ρόλο για τον οργανισμό σε όλη αυτή την υπόθεση και στο πλαίσιο αυτής της πρότασης που ασχολείται με την αξιολόγηση των τεχνολογιών για την υγεία. Ε, ευχαριστούμε. Και τώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΑ, ο κύριος, ο κύριος Ντέμερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω είναι μια χρονιά ασυνήθιστη μετά την απόφαση του Βρετανικού λαού να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα. Κατά συνέπεια, ο οργανισμός φαρμάκων πρέπει να συμμορφωθεί και να μετακινηθεί και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για τον εκτελεστικό διευθυντή και όλο το προσωπικό του οργανισμού. Από τη δική μου την ε, σκοπιά, ο κύριος Ράζη και όλοι οι συνεργάτες του έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούν για να γίνει μετακόμιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τρόπο ομαλό. Είναι σχεδόν αδύνατο βεβαίως να προβλέψουμε την κάθε μια λεπτομέρεια για το τι θα συμβεί, αλλά η πρόκληση της αλλαγής αυτής και να σκεφτούμε πώς θα επηρεάσει και την ίδια τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων είναι κάτι που το εξετάζουμε με μεγάλη προσοχή και ο Διευθυντής και ε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και προσπαθούμε να δούμε με τον καλύτερο τρόπο και από τη σκοπιά του εκτελεστικού διευθυντή τη μετακίνηση αυτή στο Άμστερνταμ και να συνεχίσουμε και το σημαντικό μα έργο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη τέθηκε ένα θέμα. Το μεγάλο πρόβλημα της αντίστασης στα αντιβιωτικά. Αυτό είναι κάτι που θα συνεχίσει να μα απασχολεί. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο. Επιτροπή. Ναι, κάποια από τα σημεία που γερθήσαν, αλλά ίσως καλύτερα να το κάνω αφού δώσει τις απαντήσεις του ο καθηγητής Ράζη. Όχι, δεν γίνεται. Τη συζήτηση θα την κλείσει ο κύριο Ράζη. Αν δεν έχετε σχόλια, πείτε το. Πολύ γρήγορα να σχολιάσω κάποια από τα σημεία που αναφέρθηκαν, κυρίως τα σημεία για την αντίσταση στα αντιβιωτικά και τις δοκιμές. Να σας καθησυχάσω να καθησυχάσω του βουλευτέ ότι η αντιμικροβιακή αντίσταση είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχει και πρόγραμμα δράση σχετικό. Το οποίο βασίζεται στην προσέγγιση για την πρόθεση της δημόσιας υγείας ε, και περιλαμβάνει πολλές πτυχές όπως την αντιμικροβιακή αντίσταση και τις σχετικές εξελίξεις στην έρευνα καθώς και την ε, έρευνα για νέα αντιβιωτικά. Ξέρετε ότι μας απασχολεί η διοδότηση των νέων φαρμάκων, νέων αντιβιωτικών, αλλά και λόγω της φύσης των αντιβιωτικών ε, πρέπει πολλές φορές να κοιτάξουμε κατά πόσο χρειάζεται ένα νέο business model και ερευνητικά ε, πρότυπα ε, για να δούμε τι μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτά. Πάντως όλα αυτά αναφέρονται κατά λεπτό στο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πίτερ. Μιας και έχουμε λίγο χρόνο, θέλω να ασκήσω για άλλη μια φορά την κριτική μου. Κύριε Ράζη, κύριε εκπρόσωπο της Κομισιόν. Προφανώς και έχουμε διαβάσει το σχέδιο δράσης και προφανώς και σας ακούσαμε πολύ προσεκτικά. Αλλά είναι επίσης προφανές ότι η Κομισιόν κάνει κάτι ελέγχους από εδώ από εκεί, μπλα μπλα μπλα. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως πριν από τον Ιούνιο του 2018 να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Εκτός αν ε, αποφασίσετε να βάλετε μπρος τις μηχανές σας. Διότι αν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, ότι δεν θα υποβάλει άλλες νομοθετικές προτάσεις από τον Ιούνιο του 2018 και έπειτα, στην παρούσα θητεία δεν θα έχουμε νομοθετική πρωτοβουλία, πρόταση, σημαίνει ότι τα επόμενα τρία χρόνια δεν θα υπάρξει τέτοια νομοθετική πρόταση. Άρα αυτό σημαίνει ότι και τα επόμενα τρία χρόνια άνθρωποι θα πεθαίνουν λόγω της μικροβικής αντιοχής. Δεν αρκεί λοιπόν το μπλα μπλα, δεν, χρεια... δεν αρκεί να συζητάμε. Από τότε που ο κύριος Ανδριοκάητης είναι Επίτροπος Υγείας, η Γενική Διεύθυνσή του δεν έχει υποβάλει ούτε μία νομοθετική πρόταση σε οποιονδήποτε τομέα. Το μόνο που, για το οποίο έχουμε συζητήσει είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, έλεος. Εγώ λοιπόν αναμένω σαφή τοποθέτηση από τον κύριο Ράζη να μου απαντήσει και να μου δηλώσει ότι δεν, υπάρχει, δεν έχουμε στη διάθεσή μας τρία χρόνια και να συμφωνήσει μαζί μου και να ασκήσει και εκείνο από την πλευρά του πίεση στην Κομισιόν προκειμένου να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Ναι, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρο. Καιρό για δράση λοιπόν. Κύριε Ράζη, έχετε το λόγο. Yeah. Ε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε, στις διάφορες ερωτήσεις και παρατηρήσεις οι οποίες βεβαίως δεν με εκπλήσουν και συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω λοιπόν. Να ξεκινήσω από το θέμα της μικροβιακής αντοχής, διότι είναι κοινή θεματική όλων των τοποθετήσεων όπως παρατήρησα σε σχέση με την AMR και το Brexit. Η μικριακή αντοχή είναι, θα παραμείνει προτεραιότητα μέχρι τελευταίας ρανίδος, για να το πω έτσι, του προγραμματισμού μας και της ε, δραστηριότητάς μας. Εγώ είμαι μικροβιολόγος ως ειδικότητα, επομένως είναι κάτι που μου είναι πολύ κοντινό όχι μόνο θεσμικά αλλά και επαγγελματικά και επιστημονικά. Πέρα από τις επίσημες δράσεις, υπάρχουν και κάποιες άλλες δράσεις που εμπίπτουν στην εντολή μας υπό την συναπόφαση και αυτές είναι ενέσεις. 2008-20 είχαμε 20 δράσεις στα κτηνιατρικά, στα της δημόσιας υγείας με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την επιτήρηση της χρήσεως των φαρμάκων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την πρωτοβουλία αυτή την ε, αναλάβαμε και προχωρεί καλώς, διότι όπως όλοι είπατε, πρόκειται για ένα εγχείρημα αρκετά περίπλοκο που περνά από διάφορα επίπεδα κίνητρα προς τους ερευνητές, προς τους παρασκευαστές, προς τους εμπορείς, αλλά ας εστιαστούμε εκεί όπου μπορούμε να έχουμε έναν αντίκτυπο, δηλαδή ο κανονισμός που θα πρέπει να διευκολύνει και να μην παρεμποδίζει αυτήν την αρκετά ήδη στενή δίωδο από την οποία διοχετεύεται όλη αυτή η προσπάθεια. Ήμασταν σε επαφή και με την FDA, την Αμερικανική, και την PMDA επίσης, διότι αν είναι να προκύψει κάτι θετικό, και ξεκινήσουν οι ρυθμιστικές αρχές μεταξύ τους να διαφωνούν, όλα αυτά θα προκαλέσουν περαιτέρω καθυστέρηση και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Γνωρίζουμε τις, ε, ότι οι κλινικές δοκιμές στο πεδίο αυτό μπορούν να επωφεληθούν τις τεχνολογίες, αλλά χρειάζεται και μία προσέγγιση προσαρμοστικότερη λέει ο μιλητής. προκειμένου να προωθήσουμε και να υποβοηθήσουμε την τεχνολογία εχμής τα θέματα EMR. Στον ΠΟΗ επίσης έχουμε πάρα πολύ καλές ε, επαφές για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την μετάβαση της γνώσεως που χρειάζεται. Επίσης με τις περιορισμένες δυνατότητες που έχουμε εντολής για τη παραμένει το θέμα στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και των ιατρών, δίνουμε και κάποιες κατευθύνσει στους κτηνιάτρους για καλύτερη χρήση των σχετικών σκευασμάτων. Είναι δύσκολο να σας πω τι θα μπορούσε να γίνει εντός ενός εξαμήνου ή μιας τριετίας, Δεν έχω πρόσθετη ενημέρωση από τους ε, εμπειρογνώμονες του ΠΟΗ ή του ΩΣΑ. Η προσπάθεια πάντως προχωρεί, καλό είναι να μην καθυστερούμε, δεν μπορώ όμως να αναφερθώ σε κάποιο συγκεκριμένο χρονοπλαίσιο. Αν έχω λίγο ακόμα χρόνο, Πρόεδρε, να περάσω σε ένα άλλο ερώτημα κλειδί. Πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα για τα εμβόλια. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των υψηλών τιμών, το οποίο είναι βεβαίως πολύ πέραν της επιρροής που μπορούμε να ασκήσουμε, αλλά κάνουμε ως συνήθως ό,τι καλύτερο μπορούμε, προκειμένου να συνεισφέρουμε στο σύνολο του πεδίου τα εξατομικευμένα φάρμακα, όπως και να θέλουμε να τα ονομάσουμε, είναι καθοδόν. Έχουμε μια διεπίπεδη προσέγγιση με έγκαιρη δέσμευση να ενημερώνουμε και να συλλέγουμε εύρωστες ενδείξεις για τη στιγμή που κάθε φάρμακο διατίθεται και προωθούμε και υποστηρίζουμε τη χρήση μητρών με έντονο, έντονη έμφαση στη συλλογή ενδείξεων γιατί είναι η μόνη προϋπόθεση για να μπορούν να εγκρίνονται τα φάρμακα αυτά, αναγνωρίζουμε βεβαίως ότι εφόσον δεν εξελιχθεί το πρότυπο τιμολόγησης θα έχουμε δυσκολίες. Θα είναι εις όλη η προσπάθεια εξυγχρονισμού που καταβάλουμε και στο επίπεδο του εξοπλισμού εφόσον δεν αναπτυχθεί μια νέα, ένα νέο σύστημα τιμολόγησης. Όπως είπα και στη σύντομη τοποθέτησή μου νωρίτερα, χαίρομαι του μέγιστου βαθμού κοινών συμβουλών, το οποίο είναι σημαντικό γιατί όταν καθόμαστε στο τραπέζι διαφαινούμε των πάντων. Αλλά εκτός διαπραγματευτικής τραπέζης υπάρχει πολύ υψηλότερο επίπεδο συνένεσης. Δεν αρκεί αυτό, αλλά είναι μια καλή αφετηρία. Εμείς συλλέγουμε την μεγάλη πλειοψηφία των δεδομένων και θα πρέπει αυτά τα δεδομένα να τα χρησιμοποιούμε όσο αποτελεσματικότερα και εκ παραλίλου γίνεται και όχι διαδοχικά δηλαδή. Από την αρχή κάθε χρήσεως, κάθε προγράμματος μπορούν και πρέπει οι φορείς να ζητούν τις ενδείξεις που έχουμε συλλέξει από την αρχή και όχι να περιμένουν όταν το πρόγραμμα είναι ήδη σε εξέλιξη. Ο συσχετισμός αποτελεσματικότητας κινδύνου είναι πάντοτε μια χρηστή ισορροπία και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. αλλά θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλους τους τομείς και την έρευνα και τον επαγγελματικό κλάδο και τους ασθενείς και την οικονομική βιωσιμότητα. Αυτό βλέπουμε περίπου σαν το δικό μας κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα, δεν ξέρω αν κάτι λησμόνησα, ελπίζω να κάλυψα τις παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα κράτη-μέλη για την ε, επικοδομητική τους κριτική και τη συνεργασία. Και ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια για το έργο του οργανισμού. Α, το, α, το, η έδρα, μάλιστα. Κοιτάξτε, η κτηριακή εγκατάσταση ε, θα πρέπει να οικοδομηθεί στο Άμστερνταμ και από ό,τι μαθαίνω το νέο κτίριο θα είναι έτοιμο τον Απρίλιο του 19 Το Νοέμβριο του 19 θα είναι έτοιμο η προσφορά του Άμστερνταμ συνοδευόταν από προσωρινή εγκατάσταση, θέμα επί του οποίου δουλεύουν δύο ομάδες, μία στην παρούσα έδρα και μία στο Άμστερνταμ, με συνεχή διεπαφή. Στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ερχόμενη Τετάρτη περιμένουμε να έχουμε τα πρώτα επίσημα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Οποιοδήποτε επόμενο βήμα μπορεί να προχωρήσει μόνον εφόσον έχουν αποσαφινιστεί όλα τα στοιχεία του προηγούμενου βήματος και δεν υπάρχει συμφωνία, λέει ο Α, μάλιστα, το χρονοπλαίσιο τώρα για τις κλινικές δοκιμές. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαφορετικό χρονοδιάγραμμα από αυτό που είχε υποβληθεί τον Ιούνιο. Παρακολουθούμε συνεχώς το θέμα και έχουμε την διαρκή στήριξη της Επιτροπής εισερχόμεθα σε μια φάση κατά την οποία η οικοδόμηση αυτών των διαφορετικών τραπεζών δεδομένων σιγά σιγά ολοκληρώνεται προκύπτει βεβαίως και μια περιπλοκότητα. Όταν κανείς προβαίνει σε δοκιμές έχουμε μια γιγαντιαία ροή δεδομένων τη μεγαλύτερη όλων των εποχών λέει ο μιλτής όπου πρέπει να έχουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο, τις ίδιες τις δοκιμές, το πλαίσιο της διαφάνειας, την προστασία δεδομένων με το σχετικό κανονισμό, την εμπιστευτικότητα των ε, εμπορικών στοιχείων. Όλα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με την κεντρική λειτουργικότητα αλλά και τη λειτουργικότητα των 28 επιμέρους συστημάτων και βεβαίως μπορεί κανείς να περιμένει να έχει ψηφιακές δυσκολίες, κάποια αισθήματα να μην ικανοποιούν τα κράτη-μέλη και τα διάφορα κράτη-μέλη όπως αντιλαμβάνεστε έχουν τελείως διαφορετικές προσδοκίες ή προθέσεις. Τώρα είμαστε αισιόδοξοι εκφύσεως λέει ο μιλητής αλλά ακόμα και όταν θα είμαστε έτοιμοι, ίσως κάποια κράτη-μέλη, ίσως πολλά κράτη-μέλη να μην είναι σε θέση να συλλέξουν, γιατί ίσως να μην συνάδουν, συνδυάζονται τα σύστημά του με την ροή δεδομένων από το κεντρικό σύστημα και μπορεί να υπάρχει και νομοθετικό πρόβλημα σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά όταν δοκιμάσουμε το σύστημα μπορεί να υποβληθούν πρόσθετες, επιβληθούν μάλλον πρόσθετες προϋποθέσεις. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς το χρονοδιάγραμμα. Περιμένουμε στις ερχόμενες εβδομάδες να έχουμε περαιτέρω διαφημίσεις για να έχουμε μια πιο ακριβή χρονική πρόβλεψη. Ευχαριστούμε, καθηγητά. Σε κάθε περίπτωση θα σας ευχηθούμε καλή τύχη. Και επειδή δεν έχουμε διάφορα, να ανακοινώσω ότι η επόμενη συνεδρία είναι στις 12 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες και σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε.